Eh, buenas tardes. Reanudamos las. Καλησπέρα σας. Ξεκινούμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Σας παρακαλώ ησυχία. Bien. A ver, Να συνεχίσουμε παρακαλώ με τη συνεδρίασή μας με το σημείο 8 της ημερησίας διάταξης. Θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Υποθέτω ότι όλοι έχετε τις κάρτες σας για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Σημείο 8. Κοινή Οργανώση Αγορών στον τομέα προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Έκθεση του κυρίου Στίβενσον. Έχουμε μία τροπολογία. Την υπαριθμόν 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ahora, ahora, ahora comienza. ¿Han votado todos? Cerramos. Για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα. Sí, han votado todos. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία από της πρότασης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή. Πάμε στο επόμενο. Κοινή ελευτική πολιτική. Τελική ψηφοφορία. Αρχή. Πέρας. Το ΕΛΚ είναι υπεράριθμο κατά έναν. Να επαναλάβουμε. A ver, repetimos, comienza la votación. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Τώρα έχει δύο υπεράριθμους στο ΕΛΚ. Βγάλετε δύο κάρτες. Σας παρακαλώ να βγάλει την κάρτα. Τώρα. Πέρας. 22 Συγγνώμη, 21 υπέρ, μία κατά. Πάμε στην επόμενη έκθεση. 10 τη ημερησία διάταξη. τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα τη ελεία και τη υγεία των ζώων λόγω τη ελίας του καθεστώτος τη Μαγιώτα τη Ένωση. Έκθεση φεραίρα. Πάμε στην τροπολογία 28. Αρχή. Τέλο. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Ε, αρχή. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 30. Συγγνώμη, ναι, 30, αρχή. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έξι Κύριε Λοβίν. Μήπως θα μπορούσαμε να δούμε τους αριθμούς στην οθόνη, γιατί δεν βλέπουμε εκεί πόσοι ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Ναι, ναι, βέβαια, να το βάλουμε. Δεν ξέρω εγώ πώς γίνεται. Αλλά όποιος ξέρει να το κάνει. Λοιπόν, ψηφίσαμε την 6. Ψηφίζουμε την 6 σε τέσσερα μέρη. Πρώτο μέρος. Πέρας. Αν δεν υπάρχει στην οθόνη, θα σας πω εγώ τα αποτελέσματα. Αν δεν ε, εμφανίσουν στην οθόνη, απορρίπτεται. 18 κατά, 3 υπέρ, 2 εποχές. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται 17 κατά, 5 υπέρ, μία αποχή. Τρίτο τμήμα, υπέρ, αυξήσει συγγνώμη, πέρας. Εγκρίνεται 13 υπέρ, 8 κατά, μία αποχή. Παρακαλώ, κυρία Άγνου. I hit the wrong button, Chairman, but it won't... Ε, κύριε Πρόεδρε, πάτησα το λάθος κουμπί, αλλά δεν έχει σημασία, το αποτέλεσμα το άκουσα. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμά του. Τέταρτο μέρο, έναρξη. Πέρα. Απορρίπτεται 18 κατά 3 υπέρ και μία εποχή. Πάμε στην τροπολογία 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 16 υπέρ 6 κατά μία εποχή. Τροπολογία 36. Αρχή. Πέρας. 16 υπέρ 5 κατά 2 εποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 38 και 7 ταυτόσιμες Ένερξη. Πέρας. Εγκρίνεται 16 υπέρ, 5 κατά 2 εποχές. Περνάμε στην τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 12 υπέρ, 9 κατά 2 εποχές. 39. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται 16 υπέρ, 5 κατά 2 εποχές. Τροπολογία 8. Α, είναι ταυτόσημη. Με συγχωρείτε με την 39. Πάμε στη 41. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ 5 κατά 2 εποχές. 42. Αρχή. Τέλος. 16 υπέρ 5 κατά 1 εποχή. Εγκρίνεται. 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16 υπέρ 4 κατά 2 αποχές. Εγκρίνεται. 48. Αρχή. Πέρας. 17 υπέρ 5 κατά 1 αποχή. Εγκρίνεται. Πάμε στην 50. Αρχή. Πέρας. 15 υπέρ, 5 κατά, 2 εποχές. Εγκρίνεται. 54. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 9 υπέρ, 12 κατά, 2 εποχές. 55. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 κατά, 9 υπέρ, 2 εποχές. 56. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται 16 πέρα 6 κατά, μία αποχή. Τροπολογία 16, ταυτόσημη με 17, 1 και 1 ρέτζι. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 16 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Περνάμε τώρα στα εκτιμώντας. Δύο. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 16 υπέρ, 5 κατά. Και βλέπετε και στην οθόνη τώρα τα νούμερα. Περνάμε στην τροπολογία 20. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 23, Ταυτόσιμο με την 3 Ρέτζι. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη. Πρέπει να ψηφίσουμε την 3. Γιατί απορρίφθηκε η 20. Την υπερθών 3. Αρχή. Τέλος. Απορρίπτεται. 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Γιατί 19 εγκρίνεται. 23 και 3 τροπολογίε. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτονται. Περνάμε στην 22. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. 5. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 26, 27 και 4. Ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Κάτι ξέχασα, λέει ο πρόεδρος. Κάποια δρομολογία ξέχασα. στη στην τροπολογία 54. Δεν ε, υπέβαλα προς ε, ψήφιση τροπολογία, γιατί νόμιζα ότι είχε εγκριθεί η τροπολογία τη Ρουινένα, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε καταρχήν. Περνάμε στην τροπολογία 14. Το βρήκατε. Να ξεκινήσουμε. Σελίδα 6. Μετά την 54 του Τυρουλιέν πάμε στην τροπολογία 14. Και στο άρθρο 6, παράγραφος 1. Εντάξει. Τροπολογία 14, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. Τώρα, ναι, 52 και 13. Αυτές καταπίπτουν. Πάμε στην νομοθετική πρόταση έτσι όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τέλος το ψήφισμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 19 υπέρ, 3 κατά και μία αποχή. Περνάμε τώρα στο σημείο 11 της μερικής διάταξης, αυτόνομες δασμολογικές ποσοστό της Ένωτης για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων αλίας στις καναρίε νήσου από το 2014 έως το 2020. Έχουν αποσυρθεί κάποιες τροπολογίες της κυρίας Πατραονέβες και την ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν κατευθείαν στο να ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα στο σύνολό του, άρχεται η ψηφοφορία. Χωρίς τροπολογίες, γιατί δεν υπήρξαν. Πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφι μία κατά, καμία αποχή. και να σημειώσουμε στα πρακτικά ότι δεν λειτουργεί το μηχάνημα της κυρίας Στομά. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκου για τον καθαρισμό ελευτικών δυνατοτήτων και χρηματική ανταπαροχή που προβλέπονται στη Συμφωνία Ελευτική Σύμπραξη μεταξύ των δύο μερών. Καταρχήν να ψηφίσουμε την τροπολογία υπερθμών 1. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Αρχή. Το κείμενο από την εισηγήτρια. Πέρας. Εγκρίνεται. 19.3. Τώρα, ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Χωρίς τροπολογίες, αρχή, πέρας. Εγκρίνεται 13 ψηφιπέρ, 8 κατά, 2 αποχές. Και τέλος, σημείο 13 πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Ακτής του Γλυφαντοστού για τον καθορισμό των ελευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη Συμφωνία Ελευτική Σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών. Τροπολογία περιθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση. Την νομοθετική πρόταση, αρχιετή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ή κονέστο. Φτάσαμε λοιπόν το τέλος των ψηφοφοριών. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. situación actual Por favor, quien se vaya a ir en silencio. Ησυχία παρακαλώ. Situación actual y perspectivas futuras Μιλάμε λοιπόν για τις μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού τομέα αλληλείας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ταϊλάνδης. Ξέρετε πως στην έκθεση αυτή, την οποία ανέλαβα εγώ, έχουμε κάνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων τον Οκτώβριο και σήμερα αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να παρουσιάσουμε την έκθεση και επίσημα. Θα λάβω λοιπόν εγώ το λόγο αμέσως και θα σας πω πως θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Γιατί ξέρω πως είναι ένα σημείο που σας ενδιαφέρει πολύ λιγότερα από τα προηγούμενα. Θα μείνουμε εμείς και εμείς, όπως συνήθως. Αυτό είναι βέβαια λυπηρό, αλλά θα περιμένουμε να βγουν οι συνάδελφοι. Και παρακαλώ όσοι αποχωρούν να μην μιλάνε. Νομίζω ότι για την έκθεση αυτή έχουμε κάνει ανταλλαγή απόψεων. Θα είμαι πολύ σύντομος και βεβαίως επιφυλάσσομαι γιατί κάποια σημεία θα μπορούσα να τα ξεκαθαρίσω αργότερα κατά τη συζήτηση. Τι θέλω να τονίσω στην έκθεση αυτή. Δεν θέλουμε να εισάγουμε ένα μεγάλο επίπεδο προστατευτισμού εδώ, γιατί δεν θα ήταν και λογικό κάτι τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για κατάργηση ε, των εμποδίων και των εισαγωγικών δασμών. Το 75% ε, του ψαριού που καταναλώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εισαγωγή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα περιοριστική στην πολιτική εισαγωγών που θα κάνουμε, απλώς θα πρέπει να, θέλ, να πιέσουμε τους εταίρους μας να είναι υπεύθυνοι. Και θα πρέπει αυτή την υπευθυνότητα να τη δείξουμε και προς τους εμπορικούς μας εταίρους και προς τις τρίτες χώρες και προς εμάς τους ιδίους. Για παράδειγμα θα πρέπει να επιδείξουμε τέτοια υπευθυνότητα προς την Ταϊλάνδη ε, στην περίπτωση που έχουμε εισαγωγές ε, αλίας, από αυτή τη χώρα είναι μια χώρα εξαγωγική και θα πρέπει να είναι βιώσιμο το εμπόριο αυτών των ειδών και να σέβεται το περιβάλλον. Και όπως πάντα να σέβεται και τα κοινωνικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή την αλληλευτική προσπάθεια και βεβαίως να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια καταπολέμησης της λαθραλίας και μια προσπάθεια να διατηρηθούν ζωντανά τα αλληλευτικά αποθέματα. Άρα λοιπόν βιωσιμότητα με την πιο ευρία ερμηνεία αυτής της ε, έννοιας. Τώρα για το προϊόν το ίδιο, τι να πω. Είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο εάν ε, εμπορευθούμε αλόγιστα μπορεί να τελειώσει. Η ζήτηση βέβαια του προϊόντας επηρεάζει τις τάσεις και στην ίδια την αλληλεία αλλά και στην εμπορία του προϊόντος. Τα ζητήματα αυτά είναι αρκετά να τα δούμε με τον τρόπο που περιγράφω στην έκθεση και νομίζω μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ευαίσθητο προϊόν το οποίο χρήζει ιδιαίτερη προστασία. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ποιος οποιαδήποτε απελευθέρωση που προσφερθεί στην Ταϊλάνδη μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα και άλλες τρίτες χώρες που εξάγουν παρόμοια προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουν ε, εισαγωγικούς δασμούς ε, ή βρίσκονται σε ένα καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι συνεκτική η πολιτική μας, η πολιτική η εμπορική, αλλά και η πολιτική αναπτυξιακή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω όπως το λέμε και στον ΠΟΕ, ελεύθερο εμπόριο, όπλο για την ανάπτυξη. Αλλά αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό που ήθελα να εξηγήσω μέσω της έκθεσής μου είναι πως για την Ταϊλάνδη δεν θέλουμε να προκρίνουμε την ανάπτυξη της χώρας μέσω μιας απελευθέρωσης της παραγωγής και της εξαγωγής αλευτικών προ... με συγχωρείτε, και δεν θα θέλαμε να οδηγήσει αυτό σε μια υπερεκμετάλλευση αυτών των πόρων. Θα πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουμε πώς θα είναι βιώσιμη η Αλία και επιπλέον πώς δεν θα κακομεταχειρίζονται τους μετανάστες οι οποίοι εργάζονται στο κλάδο σε αυτήν ε, τη χώρα. Que quede perfectamente equilibrado todo. Es decir, que se proteja lógicamente a la Unión Europea. Θα πρέπει λοιπόν να προστατευτούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά να συνδυαστούν με τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως ευαίσθητο με το δασμό ε, που επιβάλλεται αυτή τη στιγμή. Γιατί οι δασμοί, ξέρετε, μας βοηθούν και οι εξαγωγικοί και οι εισαγωγικοί να στηρίξουμε και την τοπική βιομηχανία αλλά παράλληλα να μας βοηθήσουν στο να στηρίξουμε την ανάπτυξη ε, σε κάποιες χώρες ε, που μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε στρεβλώσεις, για το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή τη στιγμή της κονσερβοποιίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε περιοχές οι οποίες εξαρτώνται από την Αλία, στη Βρετάνη, στις Αζόρες, στη χώρα των Βάσκων, στην Γαλλικία και στη Σαρδινία. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι αν κλείσουν αυτές οι βιομηχανίες θα ήταν αδύνατη η επαγγελματική επανεισδοχή των εργαζομένων και κάναμε και μία ακρόαση όχι μόνο για την εργασία των γυναικών σε αυτόν τον κλάδο και ξέρετε ότι στην περίπτωση αυτή θα μιλούσαμε για γυναίκες χαμηλής εξειδίκευσης και θα μιλούσαμε ε, για πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας που θα τίθεται σε κίνδυνο και θα ήταν δύσκολο να υπάρξει επαγγελματική επανένταξη. Έτσι λοιπόν, αυτό που ζητείτε στην έκθεση αυτή είναι η Ταϊλάνδη να σεβαστεί τους ίδιους κανόνες ανταγωνισμού που απαιτείται σε όλους τους επιχειρηματικούς φορείς του τομέα, να σέβεται το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και κλείνουμε ζητώντας το σημερινό δεσμό για τις κονσέρβες ε, ψαριού και ε, θάλασσινών που θεωρείται σε ευαίσθητα προϊόντα και να γίνονται σεβαστές οι σεβαστοί κανόνες προέλευσης χωρίς εξαίρεση. Εγώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη αυτή η έκθεση παρέχει μια καθολική προστασία και εσείς μπορέσατε να διαβάσετε και την έκθεση και του συναδέλφου Βαλέσα που νομίζω ότι είναι πολύ καλή και νομίζω ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα εργαλείο για την προστασία Τη παραγωγή και να μην δημιουργήσουμε στρεβλώσεις, κάτι που θα ήταν πολύ αρνητικό για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι σα παρουσίασα έτσι μια γενική εικόνα τη έκθεση. και τώρα είμαι ανοιχτό να ακούσω και την Κομισιόν όπως και τα σχόλια των μελών της Επιτροπής μας. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να με βοηθήσετε να βελτιώσουμε το κείμενο και σίγουρα θα είναι ευπρόσδεκτες και οι τροπολογίε αλλά και τα σχόλια. Συμφωνείτε να δώσετε το λόγο στην Κομισιόν και κατόπιν στου εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Από την πλευρά τη Κομισιόν παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος που επρόκειται να πάρει το λόγο έχει καθυστερήσει. Μήπως θα μπορούσατε να δώσετε πρώτα το λόγο στους βουλευτές. Λοιπόν, αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει να καθυστερεί η Κομισιόν. Γι' αυτό έδειξα αυτή την έκπληξη. Λοιπόν, να δώσω το λόγο του συναδέλφους πρώτα. Συνάδελφοι, είμαι εισηγητής της ΣΥΝΤΑ στο φάκελο αυτό και θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποια βασικά μηνύματα τα οποία είναι σημαντικά για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα είναι ξεκάθαρο πως βρισκόμαστε σε αμυντική ε, στάση στο θέμα αυτό και όχι μόνο για τον κορσιφιοποιημένο τόνο. Ο αποκλεισμός αυτού του προϊόντος από τις διαπραγματεύσεις δεν είναι ρεαλιστικός. Γιατί η Ταϊλάνδη έχει πάρα πολλά συμφέροντα εδώ. Η Ταϊλάνδη δεν θα δεχτεί ποτέ Αποκλεισμού τέτοιου είδου. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Κομισιόν να μεταχειριστεί τα προϊόντα αυτά ως ευαίσθητα. Δηλαδή να έχουμε ένα σύστημα ποσοστώσεων και μια κατάλληλη μεταβατική περίοδο έτσι ώστε να μην έχουμε εισαγωγές από την Ταϊλάνδη που θα δημιουργήσουν μια ανισορροπία στις ευρωπαϊκές αγορές με αρνητικές επιπτώσεις ε, και για την παραγωγή και για την ε, απασχόληση. ευαίσθητα λοιπόν προϊόντα. Μόνο αυτό είναι ρεαλιστικό. Για τους κανόνες προέλευσης, για τα μεταποιημένα προϊόντα όπως ο κονσοβιοποιημένος τόνος, στο σχέδιο γνωμοδότησης που έχω κάνει για την ίντα, προτείνω η περιφερειακή σώρευση προέλευσης να περιορίζεται στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων. Τονίζω λοιπόν ώστε να αποκλείσουμε αυτή την περιφερειακή σώρεση δεν είναι ρεαλιστικό. Γιατί η συμφωνία που έχουμε με την Ταϊλάνδη είναι ένα κομμάτι του πάζελ που στο μέλλον θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας περιφερειακής συμφωνίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, Ευρωπαϊκής Ένωσης με ΑΖΕΑΝ, μια ε, τέτοιου είδους συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Συνήθως δίνεται η δυνατότητα σόρευσης χωρών προέλευσης. Αυτό λέει ο κανόνας. Και ο στόχος εδώ είναι να προωθήσουμε την εμπορία μέσα σε εκείνη την περιοχή στην οποία δίδεται αυτή η δυνατότητα. Εγκρίθηκε αυτό πριν από ένα χρόνο σε μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής την οποία προσυπέγραψε και το Κοινοβούλιο. Ε, μία από τις χώρες που χρήζει, που, με που ευνοείται από το ε, καθεστώς, τον, το γενικό προ, προτιμησιακό καθεστώς είναι και η Ταϊλάνδη. Μπορούμε να δώσουμε μία μάχη για να περιορίσουμε τη σώρευση λοιπόν προέλευσης, αλλά δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε, γιατί κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίφαση με την εμπορική μας πολιτική. Να θυμόμαστε δε πως ό,τι και να πούμε δεν θα πρέπει να προδικάζει τη στάση που θα τηρήσει το Κοινοβούλιο στην διαδικασία ε, συμφωνίας, με συγχωρείτε συγκατάθεση, στην συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί, που θα εξαρτηθεί από το τελικό αποτέλεσμα της ε, διαπραγμάτευσης και όχι μόνο από τα όσα έχουν διαπραγματευτεί στα πλαίσια του, της Αλίας. Και τέλος, η ίντα συμμερίζεται τις ανησυχίες ε, της Επιτροπής Αλίας. Εμείς είμαστε η αρμόδια επιτροπή για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ταϊλάνδη και πολύ στενά παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις μέσω της δική μας ομάδας παρακολούθησης της χώρας. Να είστε σίγουροι πως εμείς θα σας στηρίζουμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις που αφορούν τον κλάδο της αλληλείας. Και ελπίζω, Πρόεδρε, πως θα λάβετε κι εσείς δεόντως υπόψη τις προτάσεις στην γνωμοδότηση σχετικά με τις εμπορικές πτυχές αυτού του θέματος και κυρίως ε, αυτά τα οποία μόλις έθιξα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πατράου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που ήδη ακούσαμε. Γι' αυτό ζήτησα το λόγο. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας αληθεύει ότι είναι ελληματική η Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται να εισάγει ε, ψάρια. Δεν μπορούμε όμως να διατρέξουμε τον κίνδυνο μέσω αυτών των εισαγωγών να βλάπτουμε ε, την παραγωγική μας βάση. Αυτή τη στιγμή οι εμπορικές ε, συναλλαγές με την Ταϊλάνδη ξεκάθαρα ευνοούν την Ταϊλάνδη που εξάγει την Ευρωπαϊκή Ένωση 230 τόνους ε, ε, ψαριών και παρασκευασμάτων ε, και αυτό αντιστοιχεί στην τρίτη θέση ως προς τις εξαγωγές της Ταϊλάνδης και αφήστε που η Ταϊλάνδη είναι μεγαλύτερος εξαγωγέας τόνου στον κόσμο. Κυρίως όταν μιλάμε για τις νότιες χώρες, όπως είπατε κι εσείς, είναι μεγάλος ο βιομηχανικός τομέας και τώρα με αυτήν τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Ταϊλάνδη διατρέχουμε ένα πραγματικό και σημαντικό κίνδυνο για την βιωσιμότητα του βιομηχανικού τομέα. Επιπροσθέτως, ως προς το βιομηχανικό αυτό το τομέα της Ταϊλάνδης και σε σχέση με τη συμμόρφωση με τους κανόνες, τους περιβαλλοντικούς κανόνες, τους υγειονομικούς κανόνες. ως προς ε, τις κοινωνικές συνθήκες και τις συνθήκες εργασίας, ε, ε, βλέπουμε, διαβλέπουμε και άλλους κινδύνους. Δηλαδή, διατρέχουμε κινδύνους όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και υπάρχει και άλλη διάσταση που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Οι συνθήκες παραγωγής οδηγούν σε μια τιμή κατά πολύ κατώτερη σε σχέση με την τιμή που μπορούν να προσφέρουν άλλες χώρες. Λοιπόν, μου φαίνεται ξεκάθαρο και εδώ συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι ε, ο κονσερβοποιημένος τόνος πρέπει να θεωρηθεί ε, ως ευαίσθητο προϊόν και πρέπει να ενταχθεί στη Συμφωνία Γενικευμένων Προτιμήσεων. Ε, έγραψα μία επιστολή πριν από λίγους μήνες στον Κάρολ Ντεγκούχτ εκφράζοντας ε, τις ανησυχίες μου σε σχέση με την βιωσιμότητα της ε, κονσερβοποίηση της Ευρώπης γενικότερα και των νοτίων χωρών ειδικότερα, ώστε να αναλυφθούν τα απαιτούμενα μέτρα και να αποφευθούν αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο. Ε, τους επόμενους έλαβα απάντηση από τον Επίτροπο ε, όπου ανέφερε ε, ότι γνωρίζει τον κίνδυνο που διατρέχει αυτός ο κλάδος ε, της Κονσερβοποίησης και στα πλαίσια της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου και ως προς τα υγειονομικά πρότυπα μου απήντησε ότι όντως πρέπει να συμμορφωθεί η Ταϊλάνδη βάσει και αυτών που απαιτούνται ε, δυνάμει τη κείμενη νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ένωση για το εργατικό δίκαιο και για τι περιβαλλοντικέ ε, διατάξει. Ελπίζω λοιπόν να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρξει συμμόρφωση με αυτούς ακριβούς τους κανόνες και από πλευρά της Ταϊλάνδης ε, πέραν αυτού, γιατί αυτό δεν αρκεί, πέραν αυτής της διάστασης χρειάζεται κατά προτίμηση να αποκλειστεί ο θηναλιευτικός και τομέας και τομέας κονσερβοποίησης από τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου γιατί χρειάζονται ειδικά μέτρα προστασίας. Ε, πρέπει να θεωρηθεί ως ευαίσθητο το προϊόν. Οφείλουμε να προστατεύσουμε αυτόν τον παραγωγικό τομέα. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα και στο όνομα αυτών των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου να θέσουμε εν κινδύνο ε, την ε, παραγωγική αυτή ε, βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Σύμφωνιας Ελευθέρου Εμπορίου με την Ταϊλάνδη. Οπωσδήποτε θα πρέπει να, το, να συνυπολογίσουμε και αυτή τη διάσταση και θα πρέπει να ακουστεί και η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, διότι ε, είναι και δική μας αρμοδιότητα να σταθούμε εμπόδιο σε οποιαδήποτε άλλη διαφορετική συμπεριφορά από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πλήττει την κονσερβοπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πατράου, κύριε Καρσία Γυραίο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί είναι πραγματικά καταπληκτική η έκθεσή σας και την προσυπογράφω. Εγώ τώρα τη θέση μου σε σχέση με την ε, συμφωνία δεν θα την εστιαστώ το θέμα της οικονομίας, ε, αλλά δεν μου φαίνεται ότι είναι πλέον σκόπιμες και σχετικές. Αυτό που νομίζω είναι το εξής. Δηλαδή, όχι οι κοινωνικές, όχι οι περιβαλλοντικές, ούτε οι οικονομικές ε, ε, συνθήκες, ε, ούτε οι εγγυήσει ε, των προϊόντων που εξάγονται εγγυώνται πλήρως την ποιότητα και το σεβασμό στην υγεία μας. Και εγώ δεν το πιστεύω, αλλά δεν είναι και θέμα πίστης εδώ, είναι θέμα γνώσης. Γιατί έχω συνομιλήσει με διάφορους κλάδους και με τους ακαδημαϊκούς και Όλοι γνωρίζουμε ότι ισχύουν αυτά τα πράγματα. Όμως ε, φαίνεται να είναι παράδοξο να είμαστε τόσο απαιτητικοί τη στιγμή που τα δικά μας ε, ύδατα, οι δικοί μας εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες μας ε, θα πρέπει να σέβονται συγκεκριμένε προϋποθέσεις και πολύ καλά ΜΕΛ που πρέπει να σέβονται αυτούς τους όρους και σε εργασιακό επίπεδο σε ό,τι αφορά και τις συστάσεις ε, της ΔΟΕ και θα πρέπει να σέβονται λοιπόν ε, τα δικαιώματα αυτά και θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις ποιότητας. Ε, εγώ φυσικά τα περασπίζω όλα αυτά. Αν, και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όταν μιλάμε για την αλία, μιλάμε για τρόφιμο και τελικά πρέπει να σεβαστούμε εν τέλει τον καταναλωτή, τον πολίτη που καταναλώνει τα τρόφιμα αυτά. Και τελικά εδώ μπαίνουμε σε αντιφάσεις, γιατί ε, αρνούμαστε, παραδείγματος, χάρη, να υπάρχει μια ετικέτα και στην ε, περίπτωση αυτή θα ήταν σκόπιμο να ξέρουμε σε ποια ύδατα της Ταϊλάνδη ελεύεται αυτά, από ποιε συνθήκε γίνεται η μεταποίηση, τι περιέχει αυτό το μεταποιημένο προϊόν. Μιλάμε για ε, κονσέρβες από τον θα μπορούσε λοιπόν αυτό να αποτελεί μία πρόσθετη εγγύηση όσα υπόθηκαν. Όμως νομίζω ότι τελικά αυτό που διακυβεύεται εδώ δεν ε, είναι το θέμα ε, του ότι επειδή χρειαζόμαστε τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό εισαγωγής θα πρέπει να το αποκτήσουμε από οποιαδήποτε συνθήκες. Αυτή είναι η κυρία ανησυχία δεν υπάρχουν επαρκείς εγγύησεις από τη σκοπιά, την υγειονομική και τις ποιότητες των τροφίμων. Για να αυξήσουμε το ποσοστό δεν είναι καθαρά εμπορικό το θέμα, κατά την απόψή μου. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξω γνώμη για να υποστηρίξω την πρόταση αυτή ελευθερού μπορείου ελεύθερων συναλλαγών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Γκαρσία Ιέρο, κύριος Ρωμέβα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι πολύ γενικό το σχολείο μου, κυρίως για την συμμόρφωση με τους κανόνες για την λαθραλία και την αναρχιαλία. Σε κάποιο σημείο αναφερόμαστε στον κανονισμό. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια συγκεκριμένη αναφορά στην υποχρέωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό. Υπάρχει μια διαφορά. Και επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε στη πολύ ευαίσθητη στιγμή της διαδικασίας με τους καταλόγους κτλ, νομίζω πως θα πρέπει αυτή η παραπομπή στον κανονισμό να ενισχυθεί με αυτή τη φράση. Η ε, κυρία Τωμά. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας συγχαρώ Νομίζω πως πολύ σύντομα θα έχουμε φτάσει στο τέλος και νομίζω πως αυτό που μας ζητάτε και τα όσα κάνετε εδώ περιγράφει υπέροχα τα όσα κάνουμε στην Επιτροπή μας και παίζεται η αξιοπιστία μας. Δεν μπορεί να απαιτούμε από τους Ευρωπαίους αλληλείς να σέβονται αυτά τα οποία πολύ σωστά απαιτούμε να σέβονται για το περιβάλλον, σε κοινωνικό επίπεδο, σε διατήρηση πόρων και παράλληλα να εισάγουμε προϊόντα για τα οποία δεν ισχύει καμία από αυτές τις απαιτήσει. Δηλαδή η χνηλασιμότητα, λαθραλία, υγειονομία, αμοιβαιότητα. Δεν θα σας τα αναφέρω όλα. Συμφωνώ απόλυτα με τα δικά σας συμπεράσματα, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να λέγονται ευαίσθητα τα προϊόντα αυτά, να χαρακτηριστούν και επίσης να μην προχωρήσουμε σε πλήρη απελευθέρωση από τους δασμούς. Νομίζω πως έφτασε πια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ήρθα εγκαίρω ε, για να αναφέρω την άποψη της Κομισιόν. Λέγομαι Διάννα Κόντσα, είμαι από την ΓΑΜΑ και είμαι αναπληρώτρια, επικεφαλής διαπραγματεύτρια για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταϊλάνδη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα και εγώ να παρουσιάσω κάποιες πιο γενικές πτυχές ε, της ε, συμφωνίας με την Ταϊλάνδη και εφόσον έχω την ευκαιρία θα ήθελα να κάνω μια επισκόπηση των διαπραγματεύσεων και να σας αναφέρω ποιοι είναι οι στόχοι μας με τη συμφωνία αυτή. Καταρχήν, η Ταϊλάνδη είναι πολύ σημαντική αγορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ασία μετά την Ινδονησία και η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με την Ταϊλάνδη είναι επίσης ε, ένα σημαντικό κομμάτι στο δίκτυο μας Συμφωνίων Ελευθερών Συναλλαγών ε, και θα συνεισφέρει στο να έχουμε μακροπρόθεσμα τέτοιες συμφωνίες με την ασιατική περιφέρεια. Και το 2008 το εμπόριο με την Τελάνδη έφτανε σχεδόν σε 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η τρίτος εμπορικός εταίρος για την Τελάνδη μετά την Ιαπωνία και την Κίνα με την Ταϊλάνδη θέλουμε να διαπραγματευτούμε μια νέα φιλόδοξη συμφωνία όπου θα έχουμε όχι μόνο την πρόσβαση στην αγορά για τα αγαθά αλλά και θέματα όπως ε, πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις, ε, διανοητική διοκτησία και η φόρος ανάπτυξη για να πετύχουμε μια τέτοια συνολική συμφωνία θα αποτελέσει πρόκληση. Ο κύριο στόχος είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά, στην ευρωπαϊκή αγορά για κάποια προϊόντα. Μερικά από αυτά είναι ευαίσθητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ περιλαμβάνεται και ο κοσμοπημένο τόνο. Αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν και άλλα ευαίσθητα προϊόντα για μα, όπω παραδείγματος χάρη, η ζάχαρη, το ρύζι και τα πουλερικά. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να ζητήσει από την Ταϊλάνδη πέρα από την πρόσβαση στην αγορά σε αγαθά και για μας είναι σημαντικό αυτό γιατί έχουμε αρκετά συμφέροντα όπως είναι τα αυτοκίνητα, τα αλκοολούχα ποτά και τα μεταποιημένα τρόφιμα. Όμως για μας το πιο σημαντικό τμήμα της συμφωνίας ε, είναι εκτός ε, της πρόσβασης στην αγορά για τα αγαθά, για τις υπηρεσίες, παίρνουν χάρη και για την ε, πρόσβαση στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της Ταϊλάνδης. Είναι πολύ προστατευτική η αγορά της Τελάνδης ε, και είναι πολύ διστακτική να ανοιχθούν σε ανταγωνιστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση εταιρείε που είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές συνήθως από τις τοπικές εταιρείε. Μόνο όμω ε, μια συνολική συμφωνία μπορεί να μεγιστοποιήσει τα ωφέλη για τι επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, βιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Υποστηρίζουν ε, το στόχο για φιλόδοξη συμφωνία με την Ταϊλάνδη και με τι λοιπέ χώρε στην περιφέρεια, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη αγορά για τι ευρωπαϊκέ εξαγωγέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση του του 2008 για τι διαπραγματεύσει συμφωνία ελεύθερων συνολικών με τι χώρε ΑΣΕΑΝ επίση τόνισε την ανάγκη για μια πλήρη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που θα πήγαινε πέρα από το άνοιγμα των αγορών στο εμπόριο των αγαθών. Τώρα, ο τόνος μπορεί να αποτελεί ένα σχετικά μικρό μερίδιο του εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταϊλάνδης. Είναι 1,3% της εισαγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 0,3% του συνολικού διμερούς εμπορίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε πόσο ευαίσθητο είναι το προϊόν για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα το χειριστούμε πολύ προσεκτικά την κατάλληλη στιγμή των συναλλαγών των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο. Ο τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων θα λάβει χώρα σε δύο εβδομάδες, 9 Δεκεμβρίου, και ακόμη δεν έχει υπάρξει συζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων. Αν και φυσικά γνωρίζουμε ότι ο κονσερβοποιημένος τόνος ε, είναι ένα σημαντικό συμφέρον για την ε, Ταϊλάνδη. Τα λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη αυτά, αλλά το σχέδιο έκθεσης καλεί ολικό ε, αποκλεισμό κάποιων τομέων αλλιευτικών από το άνοιγμα της αγοράς. Και να σας πω ότι είπε και ο κ. α, δεν είναι ρεαλιστικός ο συνολικός αποκλεισμό αν θέλουμε να έχουμε αυτή τη φιλόδοξη συμφωνία που σας περιέγραψα. Τώρα, αποκλεισμό ε, ενό ε, τομέα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την τελευταία οδηγήση και σε αποκλεισμού από τη δική του πλευρά και γενικά θα μειωθούν οι φιλοδοξίε. Αυτό δεν συνάδει με τι διαπραγματευτικέ οδηγίε που λάβαμε από το Συμβούλιο που ζητούν υψηλά επίπεδα φιλοδοξία και τελικά θέτουν σε κίνδυνο τη σύναψη της συμφωνίας. Από την άλλη υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι να προστατεύσουμε την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ θα δώσουμε και κάποιο άνοιγμα στους διαπραγματευτικούς εταίρους και νομίζω αυτή την οδό πρέπει να ακολουθήσουμε με τη συνεισφορά των κλάδων ε, θα εξετάσουμε τον αντίκτυπο των πιθανών παρεχωρήσεων και θα προσπαθήσουμε να εξεύρουμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της, προστασία, της προστασίας των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Μηχανίας και της προσδοκίας των Ταϊλανδών. Και σε άλλε διαπραγματεύσει, όπω με τι χώρε δεν βρήκαμε λύσει προ αυτή την κατεύθυνση και για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα. Και με αυτόν τον τρόπο σκοπεύουμε να προχωρήσουμε και με την Ταϊλάνδη είδαμε ότι ορισμένοι εκπρόσωποι της βιομηχανίας του κλάδου μας είπαν ότι η σημαντική ε, μείωση των ε, δασμών για τον κοσμοποιημένο τόνο χωρίς να πάμε σε πλήρη εξάλληψη του δασμού θα ήταν ε, μια βιώσιμη επιλογή για τον ευρωπαϊκό κλάδο. Ένα άλλο σημείο της συμφωνίας θα έχουμε ένα διμερή μηχανισμό ασφάλειας ασφαλιστικής δικλίδας, αυτός ο μηχανισμ... αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι συγκεκριμένοι ανακλάδω αλλά καλύπτουν ε, και το εμπόριο ελευτικών προϊόντων και σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις ε, όπου ε, μπορεί μια αυξημένο, αυξημένο επίπεδο εισαγωγών να έχει αρνητικές συνέπειες. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μας επιτρέψει να παρέμβουμε ταχαίως όταν ανακύψουν προβλήματα στην αγορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά πρότυπα, η Κομισιόν καλωσορίζει την ισχυρή έμφαση που δίνεται στην έκθεση για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Πράγματι, ζητάμε από τους Τελαϊνδούς μια δέσμευση να προσχωρήσουν και να εφαρμόσουν ε, τα εργατικά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ε, και τις διμερείς ε, περιβαλλοντικές συμφωνίες, ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών που λέγεται Εμπόριο και η Φόρος Ανάπτυξη. Το κεφάλαιο αυτό θα καλύψει τον αλληλευτικό τομέα και προβλέπει μεγάλη διδαρχία, όπως ο χάρη, την απαγόρευση της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας ε, και τη μη ύπαρξη διακρίσεων έναντι αλλοδαπών εργαζομένων και υπάρχει και μία αναφορά στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η, Κομισιόν, η πρόταση Κομισιόν επίσης έχει μία αναφορά σε αυτό γιατί δεν τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα και αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει πολύ μεγάλες δυσκολίες για τους Θαϊλανδούς γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα αναλάβουν ουσιαστικές δεσμεύσεις ε, με έναν το συνολικό τρόπο στην τομέα της εφορού ανάπτυξης. Άλλοι σημαντικοί στόχοι για αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για την επιβολή και τη μη παρέκκληση από την νομοθεσία την περιβαλλοντική και της ε, ε, εργασίας, όπως και διατάξεις για την εφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την καταπολέμηση της παράνομης λαφρίας και αναρχισαλίας. Επίσης, ε, θα συστήσουμε μία επιτροπή διακυβερνητική και ένα μηχανισμό να παρακολουθούμε αυτές τις δεσμεύσεις με την κοινωνία των πολιτών που θα παρακολουθεί την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού της συμφωνίας. Τα φυτογεωνομικά και γεωνομικά πρότυπα επίσης έχουν αναφερθεί και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είτε με είτε χωρίς τη συμφωνία τα εισαγόμενα προϊόντα από την Ταϊλάνδη θα πρέπει να σέβονται τους ίδιους αυστηρούς τα ίδια αυστηρά πρότυπα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν θα αλλάξει με τη συμφωνία, ακόμη και αν η συμφωνία θεσπίσει μια, ένα μηχανισμό συνεργασίας και διαβούλευσης για το θέμα αυτό, αλλά οι κανόνες παραμένουν ίδιοι και δεν θα υπάρχει παρέκκληση για κανέναν εταίρο. Και για να κλείσω, Πρόεδρο. η Ταϊλάνδη ε, είναι σημαντικός εταίρος για την κοσερβοποιημένο τόνο και διαβάσαμε πολύ προσεκτικά την ε, έκθεση και φαίνεται να δηλώνεται να δίνει την προβολική έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ταϊλάνδης και στις Εξαγωγέ τη. Όμως, σύμφωνα με τα νούμερα που έχουμε εμείς, ε, η παραγωγή της ε, Ταϊλάνδης για το μεταπημένο τόνο δεν είναι 46% αλλά μικρότερος. Και αυτό εξαρτάται με το πώς έχει γίνει ο υπολογισμός των αριθμητικών στοιχείων. Όμως να σχολιάσω και κάτι πιο μακροπρόθεσμο, μια πιο μακροπρόθεσμο προοπτική. Η θέση της Ταϊλάνδης στην παγκόσμια αγορά για το μεταπημένο τόνο μπορεί να καταστεί πιο αδύναμη τα επόμενα έτη αναμένεται πως οικονομικά στοιχεία επιτοπίου έχει ε, χτίσει την ανταγωνιστικότητά του ο τομέας στην Ταϊλάνδη μπορεί να μην διαρκέσει πολύ σε σχέση με τη συνολική μεγέθυνση της οικονομίας της Ταϊλάνδης ε, και του επίπεδου των μισθών στην Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη ήδη καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να διατηρήσει την τοπική της παραγωγή και ιδίως αναμένεται ε, μία μεγάλη ανάπτυξη στη Μιανμάρη και αυτό μάλλον θα υποσκάψει την Ταϊλάνδη. Επίσης δεν έχει εξασφαλισμένη πρόσβαση σε πρώτες ύλες η Ταϊλάνδη ενώ οι πρώτες ύλες γίνονται ο κύρια δύναμη για την βιομηχανία και για τον κλάδο και ίσως κάποιες χώρες καθεστούν πιο ανταγωνιστικές από τη Ταϊλάνδη. Όμως αυτή είναι μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική και σίγουρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η αγορά τα επόμενα έτη. Οδεύω προς το συμπερασμά μου να τονίσω ότι γνωρίζουμε ότι είναι ευαίσθητος ο τομέας του κονσερβοποιημένου τόνου. Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ευαισθησίες, τα μάλλα, αλλά και πάλι στα πλαίσια του ρεαλισμού. Και Πιστεύουμε ότι οι σημερινές, οι σύγχρονες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών ε, παρέχουν, παρέχουν τις, ε, τον καθησυχασμό που θέλετε. Για τα υπόλοιπα σημεία επίσης να σας πω ότι εργαζόμαστε με ένα διαφανή τρόπο, συζητούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με εκπροσώπους του κλάδου, έχουμε συνομιλήσει μαζί τους και θα ξαναμιλήσουμε μαζί τους και είμαι σίγουρη ότι με μια πραγματική συνεισφορά, ρεαλιστική συνεισφορά θα καταλήξουμε σε μια καλή λύση που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των διαπραγματεύσεων αυτών. Σας ευχαριστώ. Μου είπατε και εσείς κύριε Άμπο ότι εκ μέρους της Κομισιόν θέλετε να πάρετε το λόγο γιατί στις 5 κανονικά έρχεται η Επίτροπος. Δύο σημεία για την αλληλεία. Δηλαδή, εκτός από τις ε, εξηγήσεις που δόθηκαν για μια συνέπεια στα δεδομένα που υπάρχουν, Για τα υγειονομικά θέματα, να σας πω πως αρκετοί ευρωβουλευτές απαιτούν να ενταχθούν και αυτά και είναι πολύ φυσιολογικό δεν θα πρέπει τα προϊόντα που εισάγονται από την Ταϊλάνδη να θίγουν την υγεία του καταναλωτή. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Οπότε θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε πάντοτε. Για τα περιβαλλοντικά. Εδώ να υπογραμμίσω πως εδώ και χρόνια εισάγουμε συστηματικά σε τέτοιου είδους σχέσεις ένα κεφάλαιο για την <laughs> βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως ένα άρθρο για την βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων. Αν δείτε στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών που έχουμε με τη Σιγκαπούρη, θα δείτε το πιο πρόσφατο σχετικό κείμενο και είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με έναν εμπορικό εταίρο, εμπορικό εταίρο σε μια διμερή σχέση. Γιατί βέβαια πολλοί ευρωβουλευτές είπαν πως θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες. Δεν υπάρχει καλύτερος χώρος από εμπορική συμφωνία για να εφαρμοστούν τέτοιου είδους κανόνες στις πολύ πρόσφατες διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ προχωρήσαμε μια και καλύπτουμε, τουλάχιστον προσπαθούμε να καλύψουμε και τα προϊόντα καλλιέργειας. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα πάρω το λόγο εγώ στα γρήγορα για να ευχαριστήσω όσους μίλησαν. Χωρίς μικρόφωνο ο Πρόεδρος. Συμφωνώ λοιπόν, όπως και εσείς, με τις γενικές γραμμές της έκθεσης θα βελτιωθεί με τη βοήθειά σας και θα πηχήσουμε και τα όσα ακούσαμε από την Κομισιόν. Χαίρομαι που ο κύριος Βαλέσα έκανε την εκθέση στην Ίντα, γιατί είναι πολύ ευαίσθητος για τα θέματα αλίας και ξέρω πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να μας στηρίσει ενήμερους. Θα συνεργαστούμε και συμμερίζομαι με αυτόν και με κάποιον άλλον από τους προλαλήσαντες πως δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε σώρευση κανόνων προέλευσης. Για την κυρία Πατρά θα λάβουμε υπόψη τα σχολιά σας με τα οποία συμφωνούμε απόλυτα. Οι εμπορικές συναλλαγές προφανώς είναι ευνοϊκές για την Ταϊλάνδη και υπάρχουν κίνδυνοι, το έχω πει και εγώ, τους οποίους θα πρέπει να αποφύγουμε. Κυρία Ερέρο, εντάξει, η έκθεση είναι έκθεση. Νομίζω ότι καλύπτει και τις δικές σας ανησυχίες για το πώς θα εφαρμόζονται οι κανόνες. Αναμφίβολα, ναι. Όταν λέμε κανονισμός, συμμόρφωση με τον κανονισμό. Δεν νομίζω ότι εκεί μπορεί να υπάρξει διαφωνία. Και το λέω και ως εισηγητής και ως ως πρόεδρος στη μάχη για την καταπολέμηση της άναρχης και λαθρέας αλληλίας είναι ουσιαστική σημασία. Σε ευχαριστώ την κυρία Τομάς η οποία στηρίζει στο 100% τα συμπεράσματά μου Ένα σημείο το οποίο συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και το οποίο είναι σύνηθες στις συζητήσεις μας είναι οι μεγάλες απαιτήσει που βαραίνουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα και η διαφορά με τις ίδιες απαιτήσει που δεν βαραίνουν εξίσου τις, ε, τα προϊόντα τρίτων χωρών. Θα πρέπει βέβαια να είμαστε και είναι δίκαιο που είμαστε τόσο απαιτητικοί από του εαυτού μα, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε και με του εταίρου μα. Δεν μπορεί να είμαστε πολύ απαιτητικοί με τα ευρωπαϊκά προϊόντα και καθόλου απαιτητικοί με τα τρίτα. Και εδώ λέω στην Κομισιόν, όσο διευρυμένο και να είναι το πεδίο αυτών των νέων καταπληκτικών σύγχρονων συμφωνιών, θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα, κάποιο είδους προσέγγιση. Γιατί αυτή τη στιγμή οι απαιτήσει είναι τελείως διαφορετικέ στην, στην υποχρέωση συμμόρφωση με τους κανόνες για τους μεν και για τους δε. Εγώ έχω κάνει κάποιες εκτιμήσεις Δέχομαι τα όσα μου είπατε κι εσείς και δέχομαι και τα όσα είπατε για εμπορικά θέματα. Αλλά νομίζω πως θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου. Η Ταϊλάνδη είναι μια μεγάλη αγορά. Οι συμφωνίε εμπορικών ελεύθερων συναλλαγών, με συγχωρείτε, είναι πολύ σημαντικές. Είναι μεγάλος εμπορικός εταίρος. Πολύ σωστά. Και ας μιλάμε πάντα για ελεύθερη πρόσβαση προϊόν. Αλλά τότε θα πρέπει να ανοίξει και η αγορά υπηρεσιών και οι κρατικές προμήθειες. Είναι φιλόδοξη συμφωνία. Δεν έχω σε αυτό οποιαδήποτε αντίρρηση. Όμως, εάν προσθέσουμε σε αυτή τη φιλοδοξία το γεγονές πως διμερής, ε, το διμερές εμπόριο για τον τόνο είναι στο 0,8% τότε βλέπουμε μια καινούργια διάσταση. Και τι συμβαίνει με τις περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποίες έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιστούμε. Να δούμε μήπως υπάρχει κάποια συμβατότητα εδώ με τα όσα έχουμε εντάξει στη γενικότερη συμφωνία. Δεν θα πρέπει να έχουμε πλήρη αποκλεισμό. Όχι. Όταν το προτείνω είναι γιατί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Μου είπατε θα μειώσει αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας. Και πειράζει να είμαστε λίγο λιγότερο φιλόδοξοι προστατεύοντας παράλληλα την αλληλεία και την αλληλευτική βιομηχανία των συμπολιτών μας. Γιατί το ξεχνάμε. Μιλάμε για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και ξεχνάμε τους συμπολίτες μας. Και όλες αυτές οι ρήτρες διασφάλισης και τα, τα λοιπά, πολύ καλά. Αλλά τι λέμε στα ισπανικά κάλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Πολλές φορές είναι ο ίδιος ο κλάδος που πληρώνει την ύφη αυτών των συμφωνιών. Και εδώ μιλάμε για τον αλληλευτικό κλάδο. Είναι προφανές. Όταν λέτε ε, πως υπάρχουν διάφορες ε, ε, απειλές για την ανταγωνιστικότητα της Ταϊλάνδης, αν είμαστε στο 36, στο 46, εν πάση όποιο ποσοστό θέλετε, νομίζω ότι αυτή είναι απλή αριθμή. Γιατί όπως μας λένε πως εμείς δεν πρέπει να τους περιορίζουμε, είναι περίεργο πως χρησιμοποιούν το ίδιο επιχείρημα, είναι ότι αυτή τη στιγμή η θέση της Ταϊλάνδης μπορεί να αποδυναμηθεί ε, αποδυναμωθεί η Ταϊλάνδη. Ωραία, ας βάλουμε λοιπόν ρήτρες διασφάλιση για την Ταϊλάνδη, όχι για εμάς. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε αυτά τα επιχειρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε και αντίστροφα. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει την ύφη να την πληρώσει ο αλληλευτικός κλάδος. να φροντίσουμε, να προστατεύσουμε την αλληλεία μας και να έχουμε παράλληλα και μια σύγχρονη συμφωνία στα χέρια μας. Γιατί σύγχρονο είναι να προστατεύουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες. Σίγουρα υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα χρειαστεί να βελτιώσουμε και κλείνω. Είμαι ανοιχτό στο να βελτιώσω την έκθεση όσο χρειάζεται. Αλλά είμαι πεπισμένος και θα κάνω ό,τι μπορώ αυτή η συμφωνία να μην επηρεάσει αρνητικά ένα κλάδο που σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες και βεβαίως καλοδεχούμενες είναι όλες οι τροπολογίες που θα υποβάλλετε. Για να δούμε. Ήρθε η Επίτροπος. Για να δούμε λοιπόν, ξεχάσαμε κάτι στις ψηφοφορίες. Είναι για τα κοιτοειδή και την παρεπίμπτουσα αλληλεία. Εδώ είχαμε μία πρόταση για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και η διαπραγματευτική εντολή για το θέμα αυτό. Είναι κάποιες ψηφοφορίες που δεν έγινε. Προτείνω να ψηφίσουμε την απόφαση αυτή, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη διαδικασία αυτή έτσι ώστε να έχουμε σύντομα μία ε, συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δεν το ψηφίσαμε, το ξέχασα. Νομίζω ότι εδώ είμαστε αρκετοί. Υπάρχει απαρτία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Υπερψηφίζουμε. Καταψηφίζουμε. Αποχές. Άρα λοιπόν εγκρίνεται Εγκρίνεται ομόφωνα, λέει ο πρόεδρο, και λυπάμαι που το ξέχασα. Θα κλείσουμε μισό λεπτό για να δούμε αν έχει έρθει η κυρία Δαμανάκη. Α, μάλιστα, επειδή έχουμε τη διαφορά ώρα με τα Κανάρια νησιά, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Sí, he ido, rapidísimo creyendo que eran las 5 y tenía. Νόμιζα κι εγώ πω ήταν 5 και 4. Γι' αυτό έτρεχα. Δεν έχω αλλάξει το ρολόι μου. Ε, α πιούμε ένα καφέ και στι 5 κι εσείς το παθαίνετε κάμια φορά, έτσι δεν είναι. Ωραία λοιπόν, τα ξαναλέμε στι 5.